Um, Καλησπέρα, συναδελφοί. Να σας πω για το γλωσσικό καθεστώς. Υπάρχουν κάποιες γλώσσες προς τις οποίες σήμερα δεν θα υπάρχει διερμηνία, Πάντως ελληνικά μπορείτε να ακούσετε και να μιλήσετε. Επίσης, 8 ε, Νοεμβρίου το Κοινοβούλιο ε, έλαβε την ε, απόφαση η οποία τροποποιεί την 1022 και σχετικά με το καθεστώς για τις βίζες, για τις θεωρήσεις Ε, αυτή η ε, εκτελεστική πράξη ε, δημοσιεύθηκε και προωθήθηκε προς όλους τους συναδέλφους. Εάν θέλει κάποιος να αντιταχθεί σε αυτό το θέμα, παρακαλώ πολύ, πριν από τις 24 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, παρακαλώ να κοινοποιήσει αυτήν του την αντίρρηση γιατί στις 8 ε, το βράδυ 20.00 θα θεωρηθεί εγκεκριμένη. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι στις 8 σήμερα θα έχουμε ε, ψηφοφορίες, ε, να έχετε τις κάρτες σας, ε, ψηφοφορίες. Θα περάσουμε αμέσως στο σημείο 3 της εμερισίας Διάτάσταση. Ε, Έχουμε την ετήσια κατάσταση όσον αφορά ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση το 2016. Έχουμε τον κύριο Φρανκ Έγγελ, ο οποίος είναι ε, ο, είναι κεντρικός εισηγητής. 796 ήταν οι τροπολογίες οι οποίες παρουσιάστηκαν. Φρανκ, παρακαλώ, πες μας τι έχει γίνει με αυτές τις τροπολογίες. Ευχαριστώ, Κλοντ. Σωστά είπες ότι και πάλι καλά που έχουμε μονάχα 596, γιατί περίμενα πάνω από χίλιες, οπότε 596 εντάξει είναι αντιμετωπίσιμες. Έχουμε δουλέψει δε και σε συμβαστικέ τροπολογίες. Ξέρει ότι ξεκίνησα λέγοντας ότι λόγω τεχνικών ε, ε, και πολιτικών δεσμεύσεων θα ήθελα απλώς να ασχοληθώ με το κράτος δικαίου 1 και με τις ε, μεταναστευτικές ροές 2. Βεβαίως και οι περισσότερες τροπολογίες αφορούν αυτές τις δύο σημαντικές ε, τα δύο σημαντικά ε, πεδία. Ωστόσο, ήταν σαφές και για μένα ότι θα υπήρχε και πεδία προβληματισμού ε, από συναδέλφους που είχαν διαφορετική εστίαση από τη δική μου και που με κάποιο τρόπο θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η, η άποψή τους. Μιλάμε για τις μειονότητες και όσον αφορά την, τον σεξουαλικό προσανατολισμό αλλά και όσον αφορά ε, τις μειονότητες με την παραδοσιακή τους ε, μορφή. Υπάρχουν πολλές ε, προτάσεις τις οποίες ε, θα μπορούσα να λάβω υπόψη μου για τα θέματα αυτά. Επίσης, είδαμε μεγάλο προβληματισμό όσον αφορά το θέμα των παιδιών και βεβαίως και αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Υπάρχει βεβαίως κίνδυνος για πολλά ε, σημεία και στοιχεία το κείμενο να ξαναγίνει πάρα πολύ μακροσκελές. Ε, θα προσπαθήσω να το αποφύγω αυτό, ταυτόχρονα όμως προσπαθώντας ε, να βρω μια λύση για να λάβω υπόψη μου όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις στους σκιώδεις στη συνεδρίαση της ε, Τετάρτης ε, θα γίνει μια προσπάθεια έτσι ώστε ε, να βγάλουμε ίσως κάποια κομμάτια κειμένου τα οποία είναι μακροσκελή χωρίς όμως να βελτιώνουν αισθητά το κείμενο. Κύριο μέλημά μου είναι να, να παραμείνει σύντομο το κείμενο. Βεβαίως, οπωσδήποτε θα λάβω υπόψη μου όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία, γιατί κατά την άποψή μου εδώ δεν είναι πεδίο ιδεολογικής ε, αντίθεσης, ε, δεν, ε, το θέμα δεν καλεί για κάτι τέτοιο, είναι θεσμικό. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων παραμένει σε μη ικανοποιητικό επίπεδο καμία χώρα δεν ε, πέρασε από την Κρυσάρα και επομένως ε, πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη, μου, ε, μας. Αυτό ήθελα να πω και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Φρανκ. Έχουμε και κάποιους σκιώδεις. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ παρότι είναι Δευτέρα του Στρασβούργου. E ποιος θέλει να πάρει τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Κλόντο λέει η Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για τα όσα μας είπε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι εγώ ε, συμφώνησα αμέσω με το πνεύμα και την δομή της ε, έκθεσης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα για το 2016 ε, γιατί ο στόχος μας ήταν να μην έχουμε μια απλή συλλογή πληροφοριών εξ αρχής το είπαμε αυτό. Ωστόσο εγώ εκ προημίου είχα πει ότι ο συνθετικός χαρακτήρας δεν θα έπρεπε να αποβεί προζημίαν ε, της ε, ουσίας. Ε, έχουν τώρα υποβληθεί 600 τροπολογίες περίπου. Ο εισηγητής βεβαίως θα έχει την δυνατότητα μέσω ένταξης των τροπολογιών αυτών να ενδυναμώσει αυτό το κείμενο αποφεύγοντας βεβαίως τις άσκοπες και ανώφελες επαναλήψεις. Ωστόσο, κάποια στοιχεία που πρέπει να ενσωματωθούν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, ε, λαμβάνοντας ε, υπόψη και το προσχέδιο, πρέπει να δούμε αυτές που είναι προτεραιότητες και για το δικό μας, ε, για το δικό μας πολιτικό σχηματισμό. Το κράτος δικαίου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις τροπολογίες ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, τα οποία μπορούν όντως να ενδυναμώσουν το κράτος ε, δικαίου. Και όσον αφορά το άρθρο 2 των συνθήκων, αλλά και βάσει άλλων εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να υπεραμεινθούμε αυτού ακριβώς του κράτους δικαίου, ιδιαζόντως δε το άρθρο 7 και ένταξη, το δεύτερο πεδίο. Ε, κατά την άποψή μας και κατά την άποψη της ομάδας μου, ε, εδώ έχει χρησιμοποιηθεί ασαφής και όχι αρκετά καθαρή και συγκεκριμένη ορολογία. Είναι το σημείο το οποίο υπολείπεται περισσότερο ε, και κυρίως ισχολείται με την Αφρική. Εδώ μιλάμε για κράτος δικαίου εντός της Ευρωπαϊκής Επικρατείας. Οι τροπολογίες ακριβώς το τοποθετούν την μετανάστευση στο σωστό πλαίσιο, αναλύονται τα βαθύτερα αίτια, ε, ζητούνται συγκεκριμένα μέτρα από τα κράτη-μέλη, ε, γίνεται λόγος για τα στοιχεία τα οποία έχουν ελείψει έτσι ώστε να γίνει μια σωστή αντιμετώπιση και βεβαίως ε, γίνεται αναφορά σε αυτά τα βαθύτερα αίτια τα οποία σπρώχνουν κάθε μέρα τους ανθρώπους να φεύγουν από τις χώρες τους. Επίσης μέσω των τροπολογιών Λοιπόν, εγώ έχω ζητήσει ενδυνάμωση ε, ε, της προστασίας και άλλων ομάδων, όλων των ομάδων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, κυρίως δε των γυναικών και των παιδιών. Εγώ πιστεύω ότι το περιθώριο ε, ελιγμών υπάρχει και βεβαίως όπως είπατε και εσείς, τούτη τη βδομάδα θα συναντηθούμε και θα προσπαθήσουμε, τουλάχιστον εξ ονόματος της δικιάς μου πολιτικής ομάδας, εμείς είμαστε απολύτως διατεθειμένοι να ενισχύσουν ε, μέσω καρποφόρας συζήτησης ε, το προσχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, νομίζω ότι η Ναταλή από τους φιλελευθέρους θα μιλήσει εξ ονόματος της Μισελ. Ε, αντικαθιστώ τον Λουί Μισελ, ο οποίος είναι ο σκιώδης της ομάδας μας και θα προσπαθήσω να είμαι πιστή στη σκέψη του. Καταρχήν ευχαριστεί τον Φρανκ Έγγελ για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης και δέχεται πλήρως την προσέγγιση του Φρανκ έτσι ώστε η έκθεση να μην έχει ιδεολογικό περιεχόμενο καθαρά αλλά πολιτικό για να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα ως προς τα θέματα της μετανάστευσης και της διακυβέρνησης. Σε σχέση με τη διακυβέρνηση, με βάση την επικαιρότητα, θα ήταν σκόπιμο το Κοινοβούλιο να μπει σε μια συζήτηση ουσίας και ο εισηγητής να μιλήσει για μια κοινή διακυβέρνηση. Διαφορετικά θα είμαστε ένα ετερόκλητο κλαμπ όπου τα μέλη δεν συμμετέχουν, δεν τηρούν τους κανόνες του παιχνίδιου. Ως προς τα θέματα ανησυχίας, ο Λουί Μισελ θα ήθελε να ασχοληθούμε με την άνοδο του λαϊκισμού και των ακραίων τάσεων και κινημάτων σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή οικοδόμηση, κάτι το οποίο αποτελεί απειλή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό σχετίζεται και με το θέμα της διακυβέρνησης και θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα σε αυτή την έκθεση. Σύμφωνα με τον Λουί Μισελ, επίσης θεωρεί ότι κατά την κατάρτιση αυτής της ετήσιας έκθεσης και ως εισηγητής και ως Σκιώδης θεωρεί ότι γνωρίζει καταρχήν πολύ καλά ότι δεν είναι εύκολο το εγχείρημα, αλλά εμπιστεύεται τον εισηγητή για να προτείνει μια λογική και δυναμική λύση έτσι ώστε η συζήτηση μεταξύ σκιωδών να είναι ε, συνενετική. Ευχαριστούμε Ναταλή. Η ε, Λόρα Φεράρα για το EFTD. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή για το προσχέδιο που αποτελεί μια πολύ καλή βάση για την εργασία μας και εγώ ήμουνα εισηγήτρια το 13-14 για αυτή την έκθεση και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμπτύξουμε ένα τόσο ευρύ θέμα σε μια έκθεση. Υπενθυμίζω πόσο ήταν δύσκολο να φτάσουμε σε συνδυαστικέ τροπολογίες μέσα στα πλαίσια μιας σαφούς και συνεκτικής προσέγγισης. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να ορίσουμε την θεματική προτεραιότητα και να φτάσουμε σε ένα κείμενο το οποίο να είναι ευανάγνωστο. Αναφερόμαστε στο 2016 που ήταν ένα πολύ σημαντικό έτος για τις μεταναστευτικές ροές. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε το χώρο που αρμόζει σε αυτό το θέμα ως προς τις ροές. Επίσης έχουμε υποβάλει τροπολογίες για να ε, δώσουμε καλύτερη μορφή στην έκθεση και επίσης θα πρέπει να προσδώσουμε περισσότερους πόρους για να μπορέσουμε να ε, καταστήλουμε τους διακίνητες και να προτείνουμε μία εναλλακτική στην παράτυπη μετανάστευση. Και αυτό αφορά τα, τα αίτια του φαινομένου. Θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, καταστήλει οποιαδήποτε συμφωνία με δικτατορικά καθεστώτα για να μειώσουμε τις μεταστατικές ροές προς την Ευρώπη. Επίσης, η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι πολύ σημαντική. Χαίρομαι διότι ο εισηγητής ε, εισήγαγε αυτό το θέμα, το οποίο θα πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω. Ξέρουμε ότι πρόκειται για μία μάστιγα για το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να μην μειώσουμε την ποιότητα των ε, δημοσίων υπηρεσιών. Μιλάμε Μιλήσαμε για αυτό το θέμα και στην έκθεση 13-14 και χαίρομαι γιατί μας απασχολεί και στην έκθεση για το 16. Θα ήθελα η Επιτροπή να δράσει ως προς τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και για, την, για τον οργανισμό ΦΡΑ έτσι ώστε να προβούμε στην πρόληψη των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρά να βρούμε εκ των υστέρων. Υποστηρίζω λοιπόν τον εισηγητή και ελπίζω να, ότι θα τα καταφέρει και στη διαδικασία των συμβαστικών. Ευχαριστούμε Λόρα. Ο Πίτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Είμαι σίγουρος ότι είναι μια πολύ καλή αφετηρία για την συζήτηση. Καταρχήν συμφωνώ με το γεγονός ότι έθεσε στο επίκεντρο της έκθεσης το θέμα του κράτους δικαίους. Γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν ε, θεμελιώδη δικαιώματα χωρίς κράτος δικαίου. Είναι μια απαρέγκλητη προϋπόθεση. Ταυτόχρονα θα ήθελα να πω ότι εάν δούμε τις προηγούμενες εκθέσεις η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στην Ευρώπη γνωρίζει μια συνεχή επιδείνωση. Δείτε τι έγινε πριν από δύο μέρες στη Βαρσοβία όταν 60.000 διαδηλωτές άρχισαν να μιλάνε για καθαρό, καθαρή Ευρώπη και καθαρό αγνό αίμα. Ε, δεν ήταν μόνο Πολωνοί, Ούγγροι και άλλοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα ισχυρό διεθνές κίνημα της ακροδεξιάς το οποίο θα πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε γιατί πραγματικά συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε ξεκάθαρα ή να το αναφέρουμε ξεκάθαρα ε, και να το αναφέρουμε ε, είτε στο κείμενο της έκθεσης είτε μέσω τροπολογιών ότι σήμερα το πιο επικίνδυνο φαινόμενο είναι η ε, ανάπτυξη της ακροδεξιάς ε, βίας στο διεθνές σκηνικό. Ευχαριστώ, Πίτερ. Θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Φρανκ, θέλεις να απαντήσεις έχει το λόγο, ναι. Θα είμαι σύντομος, γιατί όπως είπα, θα βρεθούμε τη Τετάρτη, προκειμένου να διατρέξουμε τα θέματα, του συμβιβασμούς και θα δούμε πώς ε, θα, ποια θα είναι η αντίδραση των σκιωδών ε, ωστόσο υπάρχει ένα στενό χρονικό περιθώριο και υπάρχουν μόνο δύο μέρες μετά τα, την λήψη των ε, τροπολογιών. Εγώ θα ήθελα να είμαι έστω δυνατόν πιο ε, σαφής, περιεκτικός, αλλά και να εξαντλήσω όλο το φάσμα των θεμάτων, ε, συμπεριλαμβάνοντας το, τόσο είπε η Σεσίλ για το, την προσέγγιση στην ε, μετανάστευση. Βεβαίως ε, δεν είναι δυνατόν να τα διατυπώσουμε όλα με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και θέλουμε να, μην, ε, να συμπεριφθούν και τα στοιχεία του Λουί Μισελ όσον αφορά την έμφαση στο κράτος δικαίου. Και βεβαίως Συμφωνώ με τα όσα Λόρα σε σχέση με την ε, διαφθορά. Γι' αυτό είναι κάτι στο οποίο δεν ε, μπορούσα να επεκταθώ γιατί υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί στην έκθεση. Αλλά βεβαίως ε, η διαφθορά είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για τις κοινωνίες μας και θα έχω την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στα θέματα αυτά κάποια χρονική στιγμή. Ευχαριστώ, Φρανκ. Βεβαίω είναι πολύ δύσκολο ε, να συμπεριλάβει κανείς όλες τις πτυχέ και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω σε εσένα και του Σκιώδη για το έργο σας. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 11η Δεκεμβρίου. Είναι 8. Ε, Which item are we doing, ξέρω αν ε, μπορούμε να συμπεριλάβουμε ένα άλλο... να αναφερθούμε τώρα σε ένα άλλο θέμα τώρα. κάποιο από τα άλλα θέματα, από τα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης. Ε, το 7 που αφορά την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ε, ε, δεν θα ήθελα να κάνω τώρα την εισαγωγή, αλλά να δώσω άμεσα το λόγο στην Τζούθιτ. Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το ξέπλυμα των χρημάτων. Ε, θα έχουμε την 8η τριμερή συνάντηση αύριο στις τέσσερις. Αλλά το Συμβούλιο μου είπε ότι δεν έχουν διαπραγματευτική εντολή. Ε, υποτίθεται ότι αυτός θα ήταν, ε, αυτή θα ήταν η τελευταία ε, τριμερή συνάντηση γιατί γίνονται διαπραγματεύσεις εδώ και ένα χρόνο και βεβαίως η Μάλτα όσον αφορά την διαφάνεια τα πράγματα είναι δύσκολα ήταν δύσκολα και οι Εστονοί προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν αλλά είπαν ότι δεν είναι δυνατόν αύριο να κάνουν ε, μια συμφωνία γιατί στερούνται δεν έχουν ε, μια βάση να κινηθούν τώρα. Όσον αφορά τα ε, Paradise Papers και τις προηγούμενες διαρροές εγγράφων Παναμά και λοιπά, βλέπουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρημάτων και την ε, φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Ε, ε, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με πολιτικά δημόσια εκτεθειμένα άτομα. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη όσον αφορά κάποιου ε, οντότητε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να κάνουν κάποια πράγματα εδώ. Βλέπουμε σε αυτή την περίπτωση των Paradise ε, Papers ότι υπάρχουν εταιρείε που προσπαθούν να κινήσουν χρήματα ε, από την Ένωση εκτό και πάλι εντό και πάλι εκτό, κλπ. Και, με τώρα από αυτό δημιουργείται ένα τεράστιο παραθυράκι. Ε, δεν ξέρω Δυστυχώ, δεν μπορώ να σα πω τι θα πρέπει να κάνουμε ως επόμενο βήμα. Δεν μπόρεσα να συζητήσω με τους ε, σκιώδει. Αύριο έχει τη μια συνάντηση για τι τρει και θα δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Αλλά όπως σα είπα το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να προχωρήσει σε μια συμφωνία με εμά κάτω από το πρίσμα αυτής της πολιτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τα Paradise Papers σας ευχαριστώ πολύ. Ε, όσον αφορά το Συμβούλιο, πιστεύετε ότι όλα είναι εντάξει. Αύριο θα δούμε ποια είναι και τα αποτελέσματα. Απλώς ε, θα ήθελα να, σας, ε, να ρωτήσω τους συναδέλφους, έχετε κάτι να ρωτήσετε του, την συνάδελφο, γιατί εδώ έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, όχι από ό,τι φαίνεται. Οκ, άρα Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8. Τι να κάνουμε, να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα. Δεν νομίζω ότι έχουμε και όλους τους σκιώδεις. Is it number six? that's Mrs. Um, That's okay. No, no, I can, I can do mine quickly, if that's okay. Uh, colleagues, would you mind if I did another agenda item? Ε, σας πειράζει, συνάδελφοι, να, πάρω, να συζητήσουμε άλλο ένα σημείο της ημερησίας διατάξεως στα γρήγορα. Σημείο 5. Είναι δικό μου. Σημείο 5 της ημερησία διατάξεω. Προποθέσει εισόδου και διαμονή υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλή είναι η λεγόμενη μπλε κάρτα. Θα σας δώσω κάποιες σύντομες πληροφορίες, πολύ σύντομες πράγματι. Είμαι εισηγητής για το θέμα αυτό. 15 Ιουνίου ε, εγκρίθηκε στο, στην Κομισιόν, λίγο μετά και στο Συμβούλιο. Προχωράμε σε καλή συνεργασία με την Προεδρία και με το ε, Συμβούλιο. Τρία είναι τα ζητήματα ναι, καταλαβαίνω βεβαίω ότι αυτή η μπλε κάρτα δεν σα συγκλονίζει και δεν είναι τρομερά ενδιαφέρουσα, αλλά παρόλα αυτά μην μιλάτε πολύ. Έχουμε την εναρμόνιση των προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο είναι η ε, επέκταση του πεδίου εφαρμογής, τα θέματα τα οποία αφορούν κυρίω την διεθνή προστασία και τρίτον σε συνεργασία και με την Επιτροπή Απασχόληση τα θέματα τα οποία αφορούν αποκλειστικά την απασχόληση. Η Εστονική Προεδρία καταβάλει προσπάθειες έτσι ώστε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Βλέπω ότι ο κύριος Έγγελ που είναι ένας εκ των σκιωδών είναι εδώ, δεν βλέπω άλλους σκιώδεις. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσεις, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε όσον αφορά τον τριμερή διάλογο σχετικά με αυτές τις ειδικέ άδειε ε, ε, διαμονής. Σεσίλ για την μπλε κάρτα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, πολύ σύντομα όμως. Δουλέψαμε πολύ. Γιατί ε, πραγματικά επ' αυτού ο κανονισμός του Δουβλίνου είναι πολύ σημαντικός. Εγώ θέλω να ξέρω εάν το Συμβούλιο ε, συζητάει το σύνολο του, του, της δέσμης ε, γιατί όλα αυτά τα σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεν υπάρχει κάποιο που να είναι ελάσσονο σημασία σε σχέση με κάποιο άλλο. Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό η έγκριση να γίνει για το σύνολο της δέσμης. Ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου μπορείς να μας πεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Ευχαριστώ Σεσίλ. Ε, εδώ μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση. Η προσέγγιση και η δική μας και του Συμβουλίου είναι βάση της ε, λογικής ε, ε, της ύπαρξης νομίμων διάβλων για την ε, μεταρρύθμιση. Πρέπει να σου πω μάλιστα ότι εδώ πρόκειται για αναθεώρηση της μπλε κάρτας. Δεν είναι ε, η πρώτη νομοθεσία. Ωστόσο αυτή η μπλε κάρτα δεν χρησιμοποιείται εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, δεν χρησιμοποιείται πολύ από τα κράτη-μέλη. Οπότε μας ενδιαφέρει και ακόμα και όταν χρησιμοποιείται προκύπτουν δυσκολίες υπάρχει και ένα μέτρο όσον αφορά την εναρμόνιση ας πούμε των προγραμμάτων ε, σχετικά με ε, αυτούς που ε, έχουν δικαίωμα διεθνούς προστασίας που αποτελούν μια ειδική κατηγορία. Νομίζω πάντως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε τα μέτρα που αφορούν την νόμιμη μετανάστευση και είναι σημαντική η δουλειά και των ε, σκιωδών και τους ευχαριστώ βεβαίως για όλη τη δουλειά την οποία ε, κάνουν. Άλλες ερωτήσεις, λέει ο Πρόεδρος, για την μπλε κάρτα. Ζητώ συγγνώμη γιατί μπερδεύτηκα λίγο ή βγήκα λίγο από, την αίθουσα. Εγώ θέλω να μιλήσω για το 6, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε ακόμα στο 5, κύριε Πρόεδρε. Όντω, όντω. Ναι, λίγο μπέρδεψα την ημερήσια διάταξη. Ε, ήταν, είναι δεδαλώδηση η διαδρομή που ακολουθώ όσον αφορά την ημερήσια διάταξη σήμερα. Point, um, it is now 8 o'clock, but I've taken point And we haven't reached Πάντως ε, είμαστε στο 5 ακόμα, οπότε το 6 το οποίο σε ενδιαφέρει είναι μετά. Τώρα όμως μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, τις ε, ψηφοφορίες. Okay, colleagues, if everyone is ready, we can proceed to the vote. Ωραία, εάν είσαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Okay, and we begin with we simply have one vote. Έχουμε μία ψηφοφορία σήμερα. Η έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας 2011-93 ΕΕ για την καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της ε, παιδικής ε, πορνογραφίας. Η Άννα Μαρία Κοράτσα Μπίλντ είναι η συγγήτρια. Θέλεις το λόγο πριν ε, την ψηφοφορία, Άννα Μαρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες, όλες τις πολιτικές ομάδες, κοιόδης, βοηθούς, γιατί καταφέραμε να αποστείλουμε ένα σαφές μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα και πολύ πιο γρήγορα, έτσι ώστε να υπάρχει μηδενική ανοχή στην παιδική εκμετάλλευση και παιδική πορνογραφία. Ωραία. Τώρα περνάμε στη ψηφοφορία και αρχίζουμε με τη συμβαστική 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 52 αρχίζει ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 αρχίζει ψηφοφορία. εγκρίνεται. 54 άρχεται. Πέρας. Και εγκρίνεται. 59 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 60 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας και εγκρίνεται. Τροπολογία 68. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 69. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 70. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 71. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. 74. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 77. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 81. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 84 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 85 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 94. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 95. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 96 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 97 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 98 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 112. Άρχεται. Νομίζω είναι αρνητικό το πρόσημο που δείχνεται πέρας. Απορρίπτεται. 113. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 114 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 115 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 122 και 48 πανομοιότυπες άρχεται η ψηφοφορία. 122 και 48 από κοινού. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. εγκρίνεται. 123 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 126 και 128 πανομοιότυπες άρχεται. Πέρας. Εγκρίνονται. 133. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 144 άρχεται. Πέρας, Εγκρίνεται 145 Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 146. Άρχεται. Α, όχι, καταπίπτει. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Συμβαστική 16. 16. Συμβαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 155 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 156 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 άρχεται. Πέρας και εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Έχουμε block vote από την 1 μέχρι την 8 και την 8 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 9 άρχεται. Πέρας εγκρίνεται 10 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 12 άρχεται πέρας εγκρίνεται 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 16. Άρχεται. Το ΕΛΚ έχει έναν υπεράριθμο για τη 16 Παρακαλώ ένας να αποσύρει την κάρτα του. Θα ήθελα να το διορθώσετε. Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 17 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 19 Άρχεται. Πέρασε. Εγκρίνεται. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 25 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 26 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 27 άρχεται. Α, συγχωρείτε η 27 και 28 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνονται. 29 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 30 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 34 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 35 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τελικό κείμενο με ονομαστική η οποία και αρχίζει. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας και εγκρίνεται 46 ψήφοι υπέρ, μία κατά και μία αποχή. Να συγχαρούμε την κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία, η ώρα της ψηφοφορίας. Συνεχίζουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη και φτάνουμε αμέσως στο σημείο 6. Αγαπητοί συνάδελφοι, εάν εγκαταλείπετε την αίθουσα, παρακαλώ να το πράξετε ησύχως. Σημείο 6 Κυρία Σέπουλα, εσεί ε, παίρνετε τη θέση, αντικαθιστάτε τέλο πάντων την κυρία Φαγιόν. Of course, no problem. Birgit, are you ready? Sorry, colleagues, I'm, I'm being, trying to be helpful to everyone to finish as soon as we can. So, Λοιπόν, ε, θα πάρει το λόγο λοιπόν στη θέση της Τάνια Φαγιών. Φαγιών, who can't... Παίρνω τη θέση της κυρίας Τάνια Σφαγιών που δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Ε, πρόκειται για την ε, οδηγία σχετικά με τις ε, προϋποθέσεις. Στις 15 Ιουνίου έγινε δεκτή η πρόταση και τον Ιούλιο έγινε δεκτή και η εντολή. Στις 16 Ιουλίου πέρασε από το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να, ε, έχει, ε, να υιοθετήσει την εντολή επί του συνόλου του κειμένου για την ώρα τουλάχιστον. Έχουν μείνει ανοιχτέ κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες ε, κυρίως σχετίζονται με άλλες νομοθετικές διατάξεις και ρυθμίσεις κυρίως από τη δέσμη του ασύλου. Η κυρία Φαγιόν θα ήθελε να υπογραμμίσει ότι για την ώρα δεν έχουν υπάρξει αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, ε, ακόμα όλα βρίσκονται στον αέρα και θα εξαρτηθούν και από την ικανότητα που θα δείξει το Συμβούλιο να εγκρίνει την πλήρη εντολή. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις, έχουν γίνει δύο τριμερείς πολιτικοί διάλογοι και έχει προχωρήσει κάπως η δυνατότητα συμβιβαστικού σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε τεχνικό. Ε, οι διαπραγματευτικές ομάδες ε, ε, μπόρεσαν να συζητήσουν τα πρώτα εννέα άρθρα, συγκεκριμένα δε και το άρθρο για την εσωτερική προστασία που είναι άλλωστε και το πρώτο μείζον ζήτημα αντιπαράθεσης και προβληματίζει και τις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά όμως μέχρι το τέλος του χρόνου προβλέπονται μονάχα δύο τριμερεί διάλογοι ακόμα και είναι προφανές ότι θα ε, συνεχιστεί η προσπάθεια και με την επερχόμενη Βουλγαρική Προεδρία. Θα ήθελα να δραχθώ τι ευκαιρίες και να καλέσω το Συμβούλιο να εγκρίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, την εντολή για τι υπολοιπόμενες διατάξεις ε, του κανονισμού καθώς επίσης και να δείξει συμβιβαστική διάθεση όσον αφορά αφορά διάφορα ε, στοιχεία ε, ε, των οποίων η απόσταση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι πολύ μακρά. Θα ήθελα και ένα μικρό προσωπικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Είναι απαράδεκτο όλα τα διάφορα, όλα αυτά τα διάφορα θέματα τα οποία αφορούν την δέσμη της, του ασύλου να μην έχουν δημιουργηθεί με τρόπο συνεκτικό. Το κοινοβούλιο μας είχε την δυνατότητα να βρει μια κοινή θέση όσον αφορά πολύ ευαίσθητα θέματα, αλλά εδώ παίζουμε ποιο φταίει περισσότερο, είναι blame game. Ε, το Συμβούλιο θα πρέπει επιτέλους να έρθει με μια συγκεκριμένη θέση και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και πώς θα μπορέσουμε να πιέσουμε το Συμβούλιο έτσι ώστε να προωθήσει τις ιδέες του. Ευχαριστώ πολύ που αντικαταστήσατε την κυρία Φαγιόν ε, ενημερώνοντάς μας για, για την εξέλιξη του τριμερούς ε, διαλόγου. Και ε, συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ που περιμένατε γιατί εδώ κλείνει η συνάντηση, η συνεδρίαση ε, νομίζω ήταν πολύ έξυπνο εκ μέρους μου που έκανα τα δύο άλλα σημεία προηγουμένως διάφορα. Στι ε, στις 20 Νοεμβρίου, 21 Νοεμβρίου είναι η επόμενη συνάντηση ε, θα, θα, έχουμε και την, θα είναι κοινή με την ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ πολύ.